ασυλίας για τον κύριο Σικέρσκι στο πλαίσιο μιας οδικής ε, παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων η οποία είναι η αρμόδια από την GUE NGL